Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. First of all, I would like to... Καταρχήν, ε, έχετε τις κάρτες σας πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρία, να ρωτήσω αυτό. Εντάξει. Σε δύο λεπτά θα ξεκινήσουμε. We will start our mm, Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρείται ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο σημείο είναι ανακοινώσει τη Προέδρου. Βάσει τη γραπτή διαδικασία τη Δευτέρα και τη 8 η Οκτωβρίου, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ακυρώσουν την αποστολή στη Σουηδία που είχε προβλεφθεί να λάβει χώρα τον Νοέμβριο και να διορίσουν τον Μίχαελ Γκούσταυσον και την Edith Bauer ως ε, τακτικά μέλη του ε, Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων ε, του ΕΕ και την Πέτρα Μαϊέρ και Κότλιν Άλμπερ ως αναπληρωματικά μέλη. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ή πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Σημείο 3 της ημερησίας διάταξης, ετήσια έκθεση για τα ανθρωπινά δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Φαριά. Και θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. 8, τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, Γιατί 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε. Αλλά τι γίνεται με το μηχάνημα. Περιμένουμε τον τεχνικό. Και πάλι για την 11. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ τα αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και επειδή απορρίφθηκε η τροπολογία 5, θα ψηφίσουμε την τροπολογία 28 τρία μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Μένετε σχηρός υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. 29 καταπίπτει. 22 θα ψηφιστεί μετά την 33. Και τώρα πάμε. Τώρα πάμε στην τροπολογία 22. Τέσσερα μέρη. Πρώτο τμήμα. Τροπολογία 22, πρώτο τμήμα, υπέρ. Yes, because, ε, ε, ε, because it is in another, in another... Γιατί βρίσκεται σε άλλη παράγραφο, αλλά συμπεριλαμβάνεται σε, αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Δεν υθετήσαμε το συμβασμό, πρέπει τώρα να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 22, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Yeah, 29 falls. 29 καταπίπτει. Γιατί αθετήθηκε το 28 πρώτο τμήμα. Λυπάμαι, είναι πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκος ο κατάλογος ψηφοφοριών. Πάμε τώρα στην 22 δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 21. Ψηφίζουμε την τροπολογία 21. Υπέρ. Υπέρ για την 21. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 13 και την τροπολογία 26 ταυτόσιμες υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. Now we will vote on amendment. Ψηφίζουμε την 35. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 40. Υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά εποχές. Τώρα λειτουργεί. Για να προσπαθήσουμε. Για τη 43 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. Θα ήθελα να το επαναλάβετε την όλη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Ποια τροπολογία θέλετε. Μία προς μία. Yeah. Yes. Okay. Για να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες. Λυπάμαι που είχαμε κάποιες δυσκολίε στην αρχή. Νομίζω ότι τώρα καλά τα πάμε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται συμβαστική 9. 54 και 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 56. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά συγκρίνεται. εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 58-59 κατοπίπτουν, 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 60 σε δύο μέρη, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 Κατά αποχές συγκρίνεται Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται 79 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται Πάμε στην 81 γιατί 80 καταπίπτει. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τώρα, 85 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης, το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Συγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, congratulations. Thank you. Και τώρα σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Πρόγραμμα δικαιοσύνη. Just a moment. Just a moment. Please sit down. Μισό λεπτό παρακαλώ, καθίστε. Περιμένετε λίγο. Γιατί έχουμε και το σημείο 4. Πρέπει να ψηφίσουμε για το ημερολόγιο της Επιτροπής για το 2019. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται, τώρα μπορείτε να φύγετε. Yes. Now, uh, point five, justice program. Στο σημείο 5 είναι το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Η συγγήτρια είναι η Αγγέλικα Μίλνερ, εξέταση του σχεδίου νομοδότησης και δίνω το λόγο στην κυρία Μίλνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη να προσπαθήσω να απασχολήσω όσους από σας έχετε μείνει στην αίθουσα. Okay. Θα παρουσιάσω σύντομα το σχέδιο γνωμοδότησης για το πρόγραμμα δικαιοσύνη από το 2021 μέχρι το 2027. Τα δικαιώματα και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίζουν να ενισχύονται και να προωθούνται και να είναι κτήμα όλων των πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα προγράμματα χρηματοδότησης ε, θα βασίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες που έχουν ήδη οδηγήσει στην πρόθεση της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν όμως πολλές, πολλά κενά τα οποία παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν και νέες προκλήσεις. Από την ανάλυση μας βλέπουμε ότι δεν απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους οι πολίτες, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης. Πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν ε, περαιτέρω πρόοδοι για να μπορούν οι πολίτες να επωφελούνται από αυτές τις αξίες. Η συνεργασία, ε, η δικαστική συνεργασία σε αστικά και ποινικά θέματα δεν είναι ε, πλήρης. Το νέο πρόγραμμα δικαιοσύνη θα πρέπει να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου Δικαιοσύνη με βάση το κράτος δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την εμπιστοσύνη, ιδίως διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και προωθώντα τη δικαστική συνεργασία σε αστικέ και ποινικέ υποθέσει. Η Επιτροπή ΦΑΜ πιστεύει ότι θα πρέπει να εστιαστεί το πρόγραμμα στις εξής παραμέτρους. Να προωθήσει το κράτος δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη ε, την ε, πτυχή των γυναικών, να βελτιώσει την προσβασιμότητα στα κονδύλια και να δίνει τις ίδιες ευκαιρίες για χρηματοδότηση και τις ίδιες συνθήκες για τις οργανώσεις των πολιτών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρει κατάρτιση στους εμπλεκομένους για να βελτιώσει τη γνώση τους σχετικά με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φροντίζει ώστε να ε, παρέχεται ε, δίκαιη αντιμετώπιση και σε περιπτώσεις που επλέκονται γυναίκες ε, και παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος της γνωμοδότησής μου. Θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μλίνερ. Δίνω το λόγο στους και οδησίτες. Η κυρία Κονλιόφσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Αγγέλικα, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σημαντική γνωμοδότηση και για τις ε, προτάσεις που υπέβαλες, ούτως ώστε ε, να είναι ε, καλύτερα σε θέση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα να προωθεί τα θέματα δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χώρος της δικαιοσύνης έχει μεγάλη σημασία για την ισότητα ανδρών και γυναικών και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χωρίς να γνωρίζουμε τα θέματα δικαιοσύνης, ε, δεν θα μπορέσουμε να ε, κάνουμε πρόοδο και για την ισότητα των φύλων γενικότερα. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά ευρωπαϊκά κονδύλια για να προωθήσουμε τα θέματα της ισότητας των φύλων και τα θέματα της ε, πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε τέτοια θέματα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν χρηματοδότηση για την εκπαίδευση δικαστικών ε, εκπροσώπων και επαγγελματιών του νομικού κλάδου, όχι μόνο για τους δικηγόρους ε, και δικαστές, αλλά και για τους αστυνομικούς και άλλους ε, επαγγελματίες που πολύ συχνά είναι το πρώτο σημείο επαφής των θυμάτων βίας κατά των γυναικών. Δεν μπορούμε απλώς να υποθέσουμε ότι όλοι γνωρίζουν τα θέματα αυτά. Βλέπουμε ότι το κύριο πρόβλημα με την νομοθεσία για την ισότητα των φύλων είναι ότι δεν εφαρμόζεται επαρκώς στην πράξη. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες ε, στον τομέα ε, της δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάρτιση που θα χρηματοδοτείται ε, βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus και σύμφωνα με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποφυγή της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Στη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη, πρόσφατα είχαμε τέτοια παραδείγματα παρανόηση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και αυτό δείχνει ότι πρέπει ε, να γίνει ενημέρωση για την πραγματική έννοια των όσων ε, περιλαμβάνει η Σύμβαση για όλα τα νομικά επαγγέλματα. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες στον τομέα αυτό και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους και οδησίτες για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Νιέσκα Κογλιόφσκα. Σκιώδη εισηγήτρια Σιένα Πισιέρνα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη και την ώρα και την ε, χαμηλή παρουσία. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της για το πρόγραμμα δικαιοσύνη για την επόμενη επιτετία. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε, γιατί προφανώς το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει εγκάρσια το θέμα του φύλου και θα πρέπει φυσικά να έχει επίπτωση σε όλους τους τομείς του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Το κύριο πρόβλημα που έχουμε και αφορά αυτή την Επιτροπή και όλες εμάς είναι η πρόσβαση των γυναικών στην ίδια τη δικαιοσύνη. Ιδίως ε, όταν μιλάμε για περιπτώσεις βίας. Και εδώ οι βέλτιστες ε, πρακτικές υποστήριξης από την πλευρά των δικαστικών αρχών στην περίπτωση που έχουμε βιοπραγίες κατά των γυναικών θα πρέπει να διαδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, λοιπόν θα πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό ε, χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση δεν μπορούν να υπάρχουν και κατάλληλες πολιτικές δράσεις. Έτσι λοιπόν όλες οι δράσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις γυναίκες να καταγγείλουν τις πράξεις βίας που υφίσταται θα πρέπει να προωθηθούν. Χρειάζεται να παρακολουθήσουμε πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία παροχής βοήθειας ε, στα θύματα και πώς ε, θα εφαρμοστεί το θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος. Νομίζω ότι όλα, ελπίζω όλα αυτά να μπορέσουν ε, να ενσωματωθούν στην τελική εκδοχή του προγράμματος δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε και την έννοια της καθολικής ε, πρόσβασης στη δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και ελπίζω όλα αυτά να είναι στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος για τα επόμενα χρόνια. Τέλος, δεν έχουμε μόνο το θέμα της διάσταση του φύλου, αλλά και η ισότητα των δύο φύλων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλα τα προγράμματα και στο πρόγραμμα δικαιοσύνη. Εμείς θα συνεισφέρουμε, η δική μου πολιτική ομάδα, με κάποιες τροπολογίες στη συζήτηση για να ενισχύσουμε τη θέση της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Γυναικών. Φυσικά όλες μας εμπλεκόμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, ο κύριος Σουλέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, γιατί η διακρίση στο δικαστικό, στο δικαστικό σώμα είναι ένα από τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τις γυναίκες να έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην εξέλιξη και στην ιεραρχία. Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις, συμφωνούμε με τα σχόλια και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες για να μπει το θέμα της διάστασης του φύλου στο επίκεντρο των ε, δράσεων αυτό, αυτών. Στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι να προωθεί την εξάλληψη των διακρίσεων των διακρίσεων έναντι οποιασδήποτε, ευπαθού οποιασδήποτε ευπαθούς ομάδες όπως είναι οι μετανάστες, οι ανάπηροι και του καθεξής. Πρέπει να υπάρχει ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση και για τους δικαστές και για τους εισαγγελείς και για τους αστυνομικούς ώστε τα θύματα του τράφικινγκ και τέτοιου είδου βία προστατεύονται επαρκώ, αναγνωρίζονται, γίνονται αντικείμενα σεβασμού και δεν ε, ε, κάνει το δικαστικό ε, σύστημα μια δεύτερη θυματοποίηση του θύματος. Γιατί πολύ συχνά με αυτά που υφίσταται τα θύματα αποσύρουν τις κατηγορίες και διακόπτουν τη συνέχιση της υπόθεσης. Θα πρέπει να διαδοθεί κατάλληλο υλικό για να έχουμε την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, δεν χρησιμοποιείται αρκετά και πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω για να έχουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών, για να μπορέσουν όλοι να υποφεληθούν από αυτό και για να εξαλείψουμε τη βία με βάση το φύλλο. Τα, τα προγράμματα πρέπει να έχουν και βλέψεις για το προϋπολογισμό, να έχουν προτάσεις προϋπολογισμού συγκεκριμένες και εμείς θα έχουμε ομάδα υπερογνωμόνων, Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει ομάδα υπερογνωμόνων η οποία να εξετάζει και πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος και Θέλουμε να ε, εξετάζονται τα δεδομένα αντικειμενικά. Ευχαριστώ. Συμπεράσματα της εισηγήτριας, παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Από ό,τι άκουσα από τους κοιόδες εισηγητές, θα έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Και είναι καλό που θα ληφθεί υπόψη και από τη Βασική Επιτροπή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών, 25 Οκτωβρίου. Χαίρομαι γιατί θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ήδη είπατε εσεί ποια είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 25 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα επαναλαμβάνω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε τελειώσει. Μέχρι τις 10 συνεδριάζουμε, να ξέρετε. Αλλά βεβαίως και μπορείτε να πάτε σε άλλη συνεδρίαση αν η παρουσία σας είναι εκεί απαραίτητη. Γνωμοδότηση για το Εργαλείο Γειτονίας και Διεθνούς Συνεργασίας. Ελεονόρα Φορέντσα, εισηγήτρια. Να σας δώσω το λόγο, κυρία Φορέντσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διεθνή συνεργασία είναι ένα από του μηχανισμού που, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα που βασίζονται στην ε, υπερασπίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εδώ μιλάμε και για τα δικαιώματα των κουρτσιών και των γυναικών. Ε, μιλάμε για διάφορους ε, πολιτισμούς και τις ανταλλαγές που φέρουν αυτοί οι πολιτισμοί ο ενός στον άλλον. Αναφερόμαστε και στα δικαιώματα ε, εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για τα κρατη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουν μια συνεργασία που θα βασίζεται σε αυτές τις αξίες. Με αυτή τη βάση και με αυτή την πρόθεση εγώ κατά. Ε, το ε, πρώτο σχέδιο έκθεσης, η πρόταση κανονισμού, μηχανισμός γειτονία, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας ε, θέτει το γενικό στόχο να προωθήσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο προκειμένου να προωθήσει τους στόχους και τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ε, παρά ε, τη δήλωση αυτού του γενικού στόχου, ε, βρήκα ένα περιεχόμενο που φαίνεται να προωθεί τα συμφέροντα της Ένωσης, κυρίως ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, εις βάρος της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει πολλέ ελλείψει στο αρχικό κείμενο. Με τη στήριξη τη κοινωνία των πολιτών, αντιμετώπισα τη διεθνή συνεργασία από μια φεμινιστική σκοπιά, κάνοντα αναφορά σε όλη την πολιτική πρακτική που έχει ω στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμου. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη 5 για την ισότητα των φύλων είναι οριζόντιος και στις 17 ε, ε, διαστάσεις της Ατζέντα 23 του ΟΗΕ. Και θα ήθελα να αναφερθώ ακριβώ σε αυτό, αλλά με μια άλλη έννοια, για να αιτιολογήσω ε, κάποια μέρη αυτής τη γνωματότησης που μπορεί να μην είναι τόσο σαφή. Αναφέρομαι στις τροπολογίες 18 και 19 και στο άρθρο 9 για τις στρατικέ παρεμβάσει. Και ξεκινώ από μια προπόθεση οι γυναίκε γυναίκες ε, οι οποίες ε, ε, ε, δεν έχουν, ε, οι γυναίκες δεν έχουν φτιάξει τον πολιτισμό τους και τη λειτουργία τους βάση του εθνικισμού γιατί αγωνίζονται πάντε, πάντοτε για να καταπολεμήσουν την πατριαρχία που είναι διάχυτος σε όλους τους πολιτισμούς. Έτσι λοιπόν μέσω μιας διεθνικής κίνησης ο φεμινισμός έχει κάνει διαφορά ως στοιχείο εμπλουτισμού και γι' αυτό ως φεμινίστρες μιλάμε για τη μετανάστευση. Δεύτερον, ε, η ανταλλαγή πρακτικών ε, ε, έχει ουσιαστικά ενεργοποιήσει διάφορους αντιπαραθέσεις, αλλά ποτέ με τη μορφή πολέμου και ουσιαστικά πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα των συγκρούσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφές ότι μία φεμινιστική προοπτική και μία προοπτική δικαιοσύνης για όλους και για όλες, ο στόχος της πολιτικής συνεργασίας και ανάπτυξης ε, είναι να προστατεύσει το περιβάλλον, την παραγωγική εργασία και την αναπαραγωγική εργασία, την ασφάλεια των ανθρώπινων ζώων ε, και όχι την ασφάλεια των ε, συνόρων αυτός ο κανονισμός θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων, για την πρόθεση του διαπολιτισμικού διαλόγου, να βοηθήσει στην εξάλληψη της στόχιας, να καταπολεμήσει την ανισότητα σε κάθε της μορφή και την ε, ανισότητα μεταξύ των φύλων, να προωθήσει την ειρήνη, να ε, βοηθήσει τους πληθυσμούς ε, σε χώρες και περιοχές που υπάρχουν μεταναστευτικές πιέσεις που προκαλούνται και από φυσικές καταστροφές να υποστηρίξει μια ε, εμπορική πολιτική που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την κυρία Φορέντσα και δίνω το λόγο τώρα στους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Σολέ. Ευχαριστώ και πάλι που μου δίνετε το λόγο. Πράγματι, συμφωνώ με πολλά από αυτά που μας είπε τώρα η Ελεονόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για να καταπολεμήσει την καταστρατήγηση των, δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο και αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η Επιτροπή διάλεξε να συγχωνεύσει διάφορα εργαλεία για να δώσει περισσότερη ευελιξία. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, οι στόχοι για την ισότητα των φύλων έχουν μικρότερη ορατότητα και παίρνουν λιγότερο προπολογισμό. Αυτό συνέβη με το πρόγραμμα Δάφνη. Γι' αυτό πρέπει να διαβεβαιωθούμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι μα με τη συγχώνευση των εργαλείων αυτών. Συγχαίρω την εισηγητρία για την πρότασή τη, να υπάρχει συγκεκριμένο θεματικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων με ανεξάρτητο προπολογισμό που θα του κατακυρωθεί. Πρέπει να βεβαιωθούμε έτσι ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο και μαζί με άλλα μέτρα θα συμβάλλει για να μειωθεί η βία κατά των γυναικών, για να εξαλειφθεί, για να προστατευτούν τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα της γυναίκας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δραστών. Τέλος, Πιστεύω ότι το σχέδιο πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένε προποθέσει, όπω η αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στο φύλλο, όπω οι συγκεκριμένοι δείκτε, όπω η συλλογή ανεξάρτητων δεδομένων που έχουν να κάνουν με το φύλλο, μη σωρευμένων, μη αθρηστικών. Όλα αυτά πρέπει να λάβουν υπόψη, πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εξετάζεται το προπολογισμό. Και κάθε φορά που αποφασίζονται τέτοια προγράμματα, η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε. Επόμενη σκιώδη συγγήτρια, παρακαλώ. Εγώ ε, εκπροσωπώ εδώ τη θέση της κυρίας Μούντι, γιατί όπως είναι προφανές δεν μπόρεσε να είναι παρούσα και ζητά συγγνώμη η συνάδελφος όμως θα ήθελε να ευχαριστήσει μέσω εμπού την εισηγήτρια, την κυρία Φορέντσα, για την εξαιρετική δουλειά της επί της γνωμοδότησης αυτής για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και ως σκιώδης εισηγήτρια, η Κλέρ δέχεται θετικά ε, τα όσα λέει η εισηγήτρια για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και ε, την υποστήριξή της για την κοινότητα των ε, ΛΟΑΔΜΑ. Επίσης, ε, η αναγνώριση της όξυνσης των δράσεων κατά των οργανώσεων που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών, αναφέρεται από την κυρία Μουντή και εκτιμάται, ουσιαστικά αναφέρεται στον τεράστιο ρόλο που έχει η κοινωνία των πολιτών ε, και οι γυναικείες οργανώσεις ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και η κυρία Μούντι θα βασιστεί σε αυτές τις τροπολογίες για να ενισχύσει περαιτέρω το μήνυμα της εισηγήτριας θα επικεντρωθεί στην ένταξη της διάστασης του φύλου με την εγγύηση ότι η χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των γυναικών θα διασφαλίζεται στα εθνικά, στρατηγικά και περιφερειακά προγράμματα αλλά και στις ε, διεθνείς διαδικασίες λήψη αποφάσεων. Η κυρία Μούντι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε κυρίως στο ρόλο των γυναικών ως μία δύναμη ειρήνης και στο θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει παρουσία τους στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας μια ακόμη φορά τον αρνητικό αντίκτυπο της μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής σε γυναίκες και κορίτσια. Και πάλι ευχαριστή την εισηγήτρια και εγώ σας ευχαριστώ επίσης προσωπικά. Ευχαριστώ κύριε Πιτσέρνο. Κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. στη σημερινή συζήτηση. Σίγουρα θα υπάρχει ένας ε, καλός διάλογος ε, μεταξύ των διάφορων ομάδων βάσει του άκουσα σήμερα και σίγουρα οι τροπολογίες ε, θα έχουν στόχο να καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ευχαριστώ κυρία Φορέντσα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 26 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Σας ευχαριστώ. Στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρία μας είναι στις 8 Νοεμβρίου από τις 9 ως 12.30. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, τη Γραμματεία και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε στη συνεδρίασή μας. Καλό σας βράδυ.